Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Άρχεται η συνεδρίαση. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου και με λύπη σας πληροφορώ πως η Πίλαρ Χουάρες Μποά, η υποδιευθύντρια της